Συμβούλιο. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις εγκρίνονται. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δηλώσεις του Συμβουλίου, παρουσίαση από πλευράς του Συμβουλίου τι θέσει του αφορά το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού για το Οικονομικό έτος 2018. Παρακαλώ του ε, συναδέλφου να λάβουν υπόψη ότι για τη συζήτηση αυτή δεν προβλέπεται διαδικασία catch the eye. Δίνω το λόγο στον, Επιτρο... στον Υπουργό Κιβίνε, εκ του Συμβουλίου πρώτα απ' όλα. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να παρουσιάσω σε αυτό το Σώμα Δημοκρατίας ε, την θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2018. Έτσι όπως εγκρίθηκε αυτός από τις χώρες μέλη στις 4 Σεπτεμβρίου φέτος. Για να τηρήσω το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα είμαι συνοπτικός στις παρατηρήσεις μου. Πρώτον, Εκ μέρου του Συμβουλίου θέλω να τονίσω και να είμαι ξεκάθαρος για το γεγονό ότι το Συμβούλιο προτείνει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που τόσο στις υποχρεώσει, όσο και στις πληρωμές προτείνει αυξήσει σε σχέση με τον προπολογισμό του 2017. Και οι λεπτομέρειε έχουν ω εξή. Αύξηση 990 εκατομμύρια ευρώ, 0,6% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017 στις υποχρώσεις και στις πληρωμές. 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή 7,39% στις πληρωμές. Δεύτερον, το Συμβούλιο δίνει μεγάλη σημασία στη δημοσιονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό έχει αυξήσει τα περιθώρια πρόβλεπτων για την επόμενη χρονιά. Θέλουμε ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμό να προσφέρει ευελιξία όσο χρειάζεται. Βάσει αυτών λοιπόν, το Συμβούλιο και η Προεδρία θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα που θα μπορέσει να πάει μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο τονίζει και δαπάνες σε τομείς που έχουν μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και απορρέουν από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάπτυξη, απασχόληση, ενίσχυση της ασφάλειας και αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Οι προτεραιότητες πιστεύω ότι είναι κοινέ με αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγχρόνως, και για να τηρήσουμε τη διαδικασία του προπολογισμού έτσι όπως αυτή προβλέπεται από τις συνθήκες, το Συμβούλιο προβλέπει ότι υπάρχουν περιθώρια για εξοικονομήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση και την εκτέλεση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατόπιν τούτου, επιτρέψτε μου να μπω λίγο στο εσωτερικό του σχεδίου προπολογισμού και στις βασικές του αρχές η στήριξη της ανάπτυξη και της απασχόλησης αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητές μας. Για το 2018 θέλει το Συμβούλιο να στηρίξει ευφύ ανάπτυξη με τη συμμετοχή όλων 6,5 εκατομμύρια στι υποχρεώσει και 66,4 στι πληρωμές. 66,5-66,4. 2,1% δηλαδή και 17,5% αντίστοιχα αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2017. Όσον αφορά τώρα το 1α για την απασχόληση και την ανάπτυξη, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία που έχει αυτός ο τομέας πολιτικής, ο οποίος δείχνει καλά επίπεδα υλοποίησης. Θέλω επίσης να τονίσω και την πρόταση του Συμβουλίου για ανάπτυξη στο 1α σε σχέση με τα κριτήρια που είχαμε βάλει το 2017. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για προγράμματα όπως είναι το κόσμο, το Erasmus SIN και τον ε, πυρηνικό αφοπλισμό. Και επίσης σε τομείς όπως είναι το Horizon 2020, προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας, προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργειακά προγράμματα, οικονομική ανάκαμψη και πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Το Συμβούλιο επίσης δέχτηκε το επίπεδο υποχρεώσεων όπως προτείνεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νέες πρωτοβουλίες όπως είναι το Wi-Fi για την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή, το Σώμα Ευρωπαίων ε, Θελοντών, όπως επίσης και τα επενδυτικά σχέδια προβλέποντας ένα αποθεματικό και την επέκτασή του. Σε κάποιες γραμμές όμως του προπολογισμού, στο, στην υποκατηγορία 1α, το ποσοστό ανάπτυξης μειώθηκε εξαιτία της δυνατότητα απορρόφησης που αυτή πρέπει να είναι ρεαλιστική και δεδομένων επίση και των διοικητικών δαπανών. Για να προχωρήσουμε περισσότερο τώρα στο 1β, πολιτική συνοχή. Εδώ το βασικό στοιχείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ανάπτυξη και απασχόληση. Εδώ διατηρεί το Συμβούλιο τα επίπεδα των υποχρεώσεων έτσι όπω αυτά προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει όμω τι αιτιολογήσει να τι δει πάλι όσον αφορά τι πληρωμέ. Κυρίε και κύριοι, μια δεύτερη προτεραιότητα για το Συμβούλιο είναι να διασφαλίσει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, προστασίας και επίσης μεταναστευτικό και εξωτερικές πολιτικές. Συνεπώς, για την κατηγορία 3 όσον αφορά την ηθαγένεια, ε, δέχεται το Συμβούλιο την πρόταση της Επιτροπής για επιπλέον πόρους υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό. Το Συμβούλιο επίσης στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητοποίηση του μηχανισμού σταθερότητας που προβλέπεται βάσει της κατηγορίας αυτής. Στο 4, συνολική Ευρώπη. Ο προπολογισμό βασίζεται κατά πολύ στην πρόταση της Επιτροπής και έχει μια μείωση υποχρεώσεων ε, σε σχέση με το 2017 επειδή δόθηκαν 750 εκατομμύρια ευρώ από το κοινοτικό προπολογισμό στην διευκόλυνση για το μεταναστευτικό. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω στις κατηγορίες 2 και 5 με δύο λόγια. Στο 2 βιώσιμη ανάπτυξη και φυσική πόρη. Προτείνει κάποιε διορθώσει στο Συμβούλιο που έχουν να κάνουν με τον πρώτο πυλώνα τη κοινή γεωργική πολιτική. Οι διορθώσει έχουν ε, να κάνουν ε, βέβαια με την αναθεώρηση που θα γίνει όσον αφορά τα έσοδα και που θα συζητηθεί ε, παρετέρω το φθινόπωρο. Κάποιε εξοικονομήσεις εντοπίστηκε ότι μπορούν να γίνουν, για παράδειγμα στι εταιρικέ συμφωνίε για τη βιώσιμη αλία. Όσον αφορά το 5, δίκηση. Το Συμβούλιο μετά από λεπτομερή έλεγχο έθεσε τον προπολογισμό των κοινοτικών οργάνων σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι ένα σωστό επίπεδο, σεβόμενοι τις αρχές των οργάνων. Και έτσι καταλήξαμε σε στοχευμένες εξοικονομήσεις, φροντίζοντας για τους μισθούς και τα έξοδα τα διοικητικά όλων των οργάνων. Και υιοθετήσαμε μια δήλωση όσον αφορά τις προσπάθειες που έγιναν για να επιτευχθεί μείωση στο προσωπικό κατά 5% μέχρι το 2017 που έγινε από τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Όμως μπορεί να υπάρξουν επιπλέον βελτιώσεις για να πετύχουμε αυτό το στόχο από όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι το επίπεδο προσωπικού πρέπει να ελέγχεται συνεχώς για να διασφαλίσουμε ότι οι εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν παγιώνονται. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Θέλω να καταλήξω στο συμπέρασμά μου τονίζοντας τα Ο έλεγχος της αύξησης των δαπανών στον προπολογισμό του 2018 συγκρινόμενος με το 2017 σε τομείς που πρότεινε το Συμβούλιο θα τεθεί βέβαια στο δικό σας, ε, στη δική σας έγκριση. Υπογραμμίζουμε όμως τις βασικές αρχές των προτεραιοτήτων μας, που ήταν πρώτον μείωση της αύξησης του προπολογισμού για κάποια προγράμματα προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία στα περιθώρια, στα πλαίσια των οροφών του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεύτερον, εξοικονομήσεις στις διοικητικές δαπάνες, αντικατοπτρίζοντας όμως ε, τα προγράμματα και την ε, εκτέλεσή τους. Επιπλέον, δεν υπήρξε μείωση για την ολοκλήρωση γραμμών που προβλέπονταν για την περίοδο μέχρι το 2013 προκειμένου να πετύχει η μείωση των ε, οφειλών που είχαν συσσωρευτεί. Και δεν υπήρξε μείωση ούτε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Κατόπιν τούτο, κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συγκητές, κυρίες και κύριοι, συνδετοποιώ απόλυτα τα επόμενα βήματα που θα αναλάβουμε στη διαδικασία αυτή για την έγκριση του προπολογισμού. Περιμένω βέβαια την επόμενη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι θα εγκριθεί με το ίδιο πνεύμα με το οποίο ενέκρινε τις δικές του αποφάσεις το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ακούσατε την δική μας ε, άποψη και ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν λογικό και βιώσιμο προπολογισμό για το 2018, από τον οποίο θα μπορέσουν να υποφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Και τώρα ο Επίτροπος Έτιγκερ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Προεδρίας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, το 2018 θα είναι με δεδομένο και το προβλεπόμενο Brexit ένα κανονικό δημοσιονομικό έτος. Έχει κάνει τις προτάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα και ευχαριστούμε ιδιαίτερως γι' αυτό, έχουν διατυπωθεί οι επικοδομητικές προτάσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Οι όποιες διαφορές υπάρχουν ακόμη προς την προσέγγιση, είμαι βέβαιος πως πολύ σύντομα θα αντιμετωπιστούν με ένα, και θα καταλήξουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Στην, στο υπόβαθρο του, του προϋπολογισμού δεν έχουμε διαφορές, ούτε στους στόχους που επιδιώκουμε. Με την ίδια αποφασιστικότητα λοιπόν επιδιώκουμε την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, την συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών και με οικονομικά μέσα, την ενίσχυση της ασφάλειας προς το συμφέρον των πολιτών και την εξασφάλιση της σε υψηλό επίπεδο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ε, διοικητικά κονδύλια, στις ταπάνες για το προσωπικό και τη λειτουργία έχουν ε, συμπεριλάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες οικονομίες και μέσα στο στόχο του 5% έχουμε ε, ακολουθήσει τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Η πρόταση τώρα του Συμβουλίου αναφέρεται σε 1,5% επιπλέον περικοπή στις δαπάνες. Εδώ έχουμε επιφυλάξει και ανησυχία για το κατά πόσο μπορούμε αυτό να το επιτύχουμε, διότι αν μειώσουμε ακόμη περισσότερο το προσωπικό μας, οι υπηρεσίες μας και η δυνατότητα επιτέλεσης του έργου τους ε, τίθενται σε κίνδυνο. Για τα προγράμματα συνοχής. Και το 2018 συνεχίζουμε με τα προγράμματα συνοχής χωρίς αλλαγές, με ε, λειτουργία τους σε ρυθμούς καλούς. Υπάρχουν μέχρι τώρα, ε, έχουν σημειωθεί κάποιες καθυστερήσεις. Ε, μπορέσαμε χάρη στη συγχρηματοδότηση να απεμπλέξουμε ορισμένα έργα που είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα και πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση για του χρόνου να έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και να μην έχουμε εκκρεμείς λογαριασμούς στις Βρυξέλλες γιατί έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση και ως προς τους μη εξοφληθέντες ε, λογαριασμούς ναι. και σε αυτό θα χρειαστεί ε, να πείσουμε και τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στην ε, αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Επίσης, το Wi-Fi for Europe αλλά και άλλα σημαντικά προγράμματα έχουν τύχει και ευχαριστούμε γι' αυτό της υποστήριξης και του Συμβουλίου. Είναι σε μια φάση αρχική και χρειάζονται την υποστήριξη και την οικονομική και τη χρηματοδότησή τους. Οι συνομιλίες στον τριμερή διάλογο του τις επόμενες εβδομάδες θα αξιοποιηθούν, ε, θέλω να επισημάνω, ώστε να κοιτάξουμε ιδιαίτερα τους τομείς ε, του μέλλοντος, ε, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας για τα επόμενα χρόνια. Μας ανησυχούν δηλαδή οι περικοπές στον ορίζοντα 2020 κατά ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί και τα τρία θεσμικά όργανα το 3% του ε, κοινού μας ΑΕΠ να αφιερώνεται στην έρευνα και την καινοτομία. Τώρα είμαστε στο 2% μόνο. Όσο λιγότερο λοιπόν προσφέρουμε στο στόχο αυτό, τόσο χειρότερη είναι χειρότερα τα επίπεδα της επίτευξής του. Θα πρέπει κάθε χρόνο ως Ευρωπαίοι να ε, επενδύουμε 150 δισεκατομμύρια ευρώ στο στόχο αυτό. Τώρα το να περικόψουμε κατά 500 εκατομμύρια τη χρηματοδότηση που έχουμε τώρα εξασφαλίσει είναι λάθος μήνυμα και μην λησμονούμε ότι υπάρχει πολύ σημαντική προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Ε, επί παραδείγματι, ύστερα από τις ε, περικοπές στα τομέα της ψηφιακής ε, τεχνολογίας κινδυνεύουμε να χάσουμε τρία από τα τέσσερα μεγάλα συμβόλαια ε, και έτσι ε, υπολοιπόμαστε πολύ και της Silicon Valley και της Κίνας και μεγάλων άλλων ανταγωνιστών. Το ίδιο και στην έρευνα για τον καρκίνο, για τις μεγάλες αρρώστιες, για την προσωποποιημένη ιατρική περίθαλψη θα καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο σχέση με τους ανταγωνιστές μας η κβαντική τεχνολογία που μας είχε απασχολήσει και στα προηγούμενα μου καθήκοντα όπου έχουμε αναπτύξει πρωτοπόρες πρωτοβουλίες με πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες τις οποίες συμμετέχουν ε, Ινστιτούτα ερευνητικά, κράτη, πανεπιστήμια ε, το να δει αυτό περικοπή, περικοπές και κυρίως τη στιγμή όπου επενδύουν η Google, η Amazon, η Yahoo ε, η Microsoft δισεκατομμύρια στον ίδιο τομέα είναι πολύ εσφαλμένο μήνυμα. Δεν κάνουμε μια ε, σύγκριση θεωρητική. Δεν είμαστε ένα θεωρητικό ανταγωνισμό, αλλά ένα πολύ πραγματικό ανταγωνισμό και προσπαθούμε να σας πείσουμε για τη σημασία των έργων αυτών και για τη σημασία των, και τις συνέπειες των περικοπών που θα οδηγήσουν και σε κατάργηση κάποιων προγραμμάτων. Η πρωτοβουλία για το συνδε, την Ευρώπη, το ΙΤΕΡ, το Κοπέρνικους, το Γαλιλαίος δεν μπορούν να δουν περικοπή. Ε, κονδυλίων διότι θα πάψουν να λειτουργούν σε λίγο. Εάν δεν επενδύσουμε τώρα θα πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερα το 2020-2022 για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος τώρα. Λοιπόν πρέπει να δεσμεύσουμε ή ακόμα να συγκρατήσουμε δηλαδή αλλά και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη χρηματοδοτική μας πρόβλεψη έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τρέχουμε πίσω από την πρόοδο που θα έχουν επιτύχει άλλοι οι Αμερικανοί, οι Ασιάτες. Και βεβαίως το θέμα της ασφάλειας και των αισθανευτικών ροών ε, πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με μεταγνώσεως λόγου να μιλήσουμε για το αν υπάρχουν δυνατότητε για περικοπές κονδυλίων ή τι συνέπειε μπορεί να έχουν αυτές. Το 2018 είναι δυνατόν να βρεθεί μια ε, λύση συμβαστική εάν μπορέσουμε αυτά τα θέματα να τα λύσουμε και ίσως μπορέσουμε και να μην εξαντλήσουμε όλο το χρόνο που έχουμε σε συνεδριάσεις προβλέψει για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μπορούμε δηλαδή με μια μικρή προσπάθεια να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να ε, έχουμε έναν καλό προπολογισμό για το 2018. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, προσβλέπω σε πολύ καλή συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου αλλά και με τους ηγητές του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο και τώρα λαμβάνει το λόγο ο Επίτροπος, ε, Κύριος Μούρης, ανησυχητής, παρακαλώ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ε, κύριε εκπρόσωπε της Ιστονικής Προεδρίας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, μπαίνουμε σε μια αποφασιστική φάση σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2018. Έχουμε περάσει το πρώτο μέρο ε, του 2017 για να συμφωνήσουμε για τι πολιτικέ προτεραιότητε. Και αυτό το κάναμε ε, με επιτυχία. Είπαμε ότι η απασχόληση, η ανάπτυξη, η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να είναι οι πολιτικέ προτεραιότητε του προπολογισμού τη Ένωση για το επόμενο έτο. Αυτέ είναι οι σωστέ προτεραιότητε, διότι αυτό απαιτούν, αυτό περιμένουν οι πολίτε από την Ευρώπη. Και εκεί είναι και η αξία τη Ευρώπη. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει οι υποσχέσει ε, που δώσαμε στι αρχέ του έτου ε, να τηρηθούν. Δεν είναι αξιόπιστο το να πούμε ότι θέλουμε μια πιο καινοτόμη Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να περικόπτουμε 591 εκατομμύρια ευρώ από την κοινοτομία και τα προγράμματα έρευνας. Δεν είμαστε αξιόπιστοι όταν λέμε ότι θέλουμε υποδομές στην Ευρώπη και βελτίωσή τους, ε, ψηφιακή ε, δρόμοι, ε, σιδηρόδρομοι και κόβουμε πολύ σημαντικά ποσά από μεγάλα project ε, ε, υποδομών και από, το και από την ψηφιακή Ευρώπη. 1,7 ε, δις είναι οι περικοπέ και είναι μεγάλο το ποσό. Αυτό που προτείνει το Συμβούλιο είναι ένα προπολογισμό για μια πιο αδύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι λιγότερε επενδύσει σήμερα σημαίνει μια πιο αδύναμη Ευρωπαϊκή Οικονομία στο μέλλον. Η Επιτροπή το είπε αυτό, έδωσε παραδείγματα πολύ πιστικά από τον ψηφιακό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε στο πρώτο ε, εξάμεινο ότι η απασχόληση, η ανάπτυξη, η ασφάλεια πρέπει να είναι προτεραιότητες μας και έχει προετοιμάσει έναν προπολογισμό εξαιρετικά καλό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα ε, του περισσότερου πόρου που έχουμε ε, για, την έρευνα, τις, τα σχέδια υποδομών, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, να είμαστε δίπλα στου γεωργού, ιδιαίτερα στου νέου γεωργού και θα πρέπει ε, να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας ό,τι αφορά την συνοχή και τα διευθυντικά ταμεία. Ε, τα χαμηλά ποσοστά απορρόφησης στο πρώτο εξάμεινο δεν σημαίνει ότι θα μείνουν χαμηλά και στα επόμενα έτη. Ε, αντιθέτως, τα project ε, σιγά σιγά ε, θα επιταχυνθούν και θα χρειαστούν τα χρήματα αυτά τα ερχόμενα έτη. Είναι ένα πολύ κακό μήνυμα ε, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους πολίτες, προς ΜΚΟ το να μην πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους λογαριασμούς της. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από όλους τις επόμενες εβδομάδες να συναντηθούν για να φτάσουμε σε έναν καλό προεπολογισμό το 2008 για την Ένωση που να βασίζεται στις επενδύσεις, στην υποστήριξη της έρευνας, της κοινοτομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαντικά project, ε, χρήματα δηλαδή διατεθούν για τα καλά αυτά project που έχουν. Να είμαστε κοντά ε, στην γειτονία μας, στις γειτονικέ μας χώρες, στον Νότο, στην Ανατολή, να βελτιώσουμε την ασφάλεια, να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες, ε, του οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχουν για να βελτιωθεί η ασφάλεια των πολιτών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο έτερος εισηγητής, κύριος Σάσχουρθ, τρία λεπτά επίσης. Uh, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τον Απρίλιο φέτος ε, συμφωνήσαμε να αυξηθεί ο ετήσιος της Ένωσης ε, κατά 3,2%. Λαμβάνοντας υπόψη το ποστό της, ε, του πληθωρισμού, ήταν μια ρεαλιστική πρόταση αυτή και θα πρέπει να είναι ένα benchmark και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να πω σήμερα ότι η πλειοψηφία των άλλων θεσμικών οργάνων το δέχονται αυτό και έχουν υποβάλει παρεμφερείς προτάσεις. Υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων ε, της έχει ζητηθεί να ε, αυξήσει τις δραστηριότητε του, οπότε αυτό σημαίνει και μια αύξηση των δαπανών σημαντική και αντίστοιχη. Επίσης, το Ελληνικό Συνέδριο έχει αυξήσει το φόρτο εργασία του και εκεί δέχομαι ότι είναι θεμητό, είναι λογικό να ζητηθεί αύξηση του προπολογισμού. Και τρίτον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εδώ και καιρό ζητάει αύξηση του προπολογισμού, είναι πιο μεγάλο το κόστος μετάφρασης, είναι πιο πολλές οι υποθέσει. υπάρχουν και πολύ σημαντικά ζητήματα ασφάλεια που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο δικαστήριο. Ε, αυτό το επιπλέον κόστο βέβαια μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο έχει περικόψει υπερβολικά σε κάποιους άλλους τομείς. Πρέπει κάποια από αυτά τα επίπεδα να επανέλθουν. Όμως ε, για να παραμείνουν, να παραμείνει το σύνολο των δαπανών υπό έλεγχο πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εξοικονόμηση. Εγώ πρότεινα αυτό το επιπλέον κόστος να καλυφθεί μέσω κέρδος, κέρδος επίπεδο αποτελεσματικότητας και το συνέδριο ε, ως ένα βαθμό ακολούθησε αυτήν την ιδέα. Από την άλλη θα πρέπει να υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία και αναδιανομή της χρηματοδότησης. Προτείνω λοιπόν να παγώσουμε τον προπολογισμό του Ελληνικού Συνετού, του Επιτροπής των Περιφερειών και της ΕΟΚΕ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνική Επιτροπή, για το 2018. Επίσης, βεβαίως, γνωρίζω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, βλέπει το κόστος της να αυξάνεται. Αυτό έχει να κάνει με την, το αυξημένο, προσω... τον αυξημένο αριθμό ατόμων που εργάζονται εκεί, αλλά και λόγω των προγραμμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αυτού πρέπει να απορροφηθεί από τον παρόν προπολογισμό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Μπορώ να δεχτώ ότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή προς τα πάνω όταν θα έχουμε τα ακριβή στοιχεία. Πρόεδρε, ε, σας ζητώ να λάβετε υπόψη ότι αν συμφωνείτε μαζί μου ότι το 2,3% είναι ένα λογικό ποσοστό, είναι μια λογική αύξηση του προπολογισμού, εάν θέλουμε να το εφαρμόσουμε αυτό και στις λοιπές κατηγορίες, θα πρέπει να παρθούν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Εγώ είμαι διατεθειμένος να συζητήσω το, ζήτημα αυτό και τις προτάσεις μου με τους κυρίως συζητητές και να, ελπίζω να λάβω την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Άσφερ. Το λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών, ο κύριος Αρτουή. Αλλά δεν τον βλέπω στο ημικύκλιο. Οπότε ο Υπουργός ε, Κιδίνε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας που ήταν γεμάτες πάθος και ενθουσιασμό. Επιτρέψτε μου να απαντήσω με λίγα λόγια. Κύριε Επίτροπε, αυτό που είπατε, κυρίως για την έρευνα, όντως είναι πολύ σημαντικό και να ξέρετε ότι το Συμβούλιο το αντιμετωπίζει θετικά. Θα το επαναφέρουμε στο συναδέλφο στο Συμβούλιο και είμαι σίγουρος ότι θα το συζητήσουμε σε βάθος στη διαδικασία αυτή προπολογισμού. Είναι πολύ καλό αυτό που είπατε και αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό, να το συζητήσουμε, να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή την μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Επίρου μας. Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ πολύ και όλους σας για τόσο μας είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες και αυτά. Ε, μπορώ και υπόσχομαι ότι θα τα συζητήσω με τους συναδέρφους και ξανά με σας πολύ σύντομα όταν θα περάσουμε στις συζητήσεις σε βάθος για τον προπολογισμό αυτών. Κύριε Άσουερτ, και σας σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Είναι ε, πολύ καλά τα όσα θέσατε και αυτά θα τα υπόψη μας στην ε, εξέταση του προπολογισμού που θα συνεχιστεί όταν ε, φτάσουμε στο θέμα του διοικητικού κόστους. Κατόπιν τούτον όμως και αναγνωρίζοντας ότι μπαίνουμε στη διαδικασία των τριμερών διαλόγων. Θέλω να τελειώσουμε τη σημερινή συζήτηση με κάποιες ακόμα παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, εννοείται σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Συμβουλίου, εκ μέρους ε, του εαυτού μου του ίδιου και των συναδέρφων και σας ε, ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε τόσο νυχτά και με τέτοια ειλικρίνεια τις παρατηρήσεις σας. Για μένα η σημερινή συζήτηση έδειξε ότι όλοι θέλουμε να αγωνιστούμε για το κοινό καλό και να πετύχουμε το καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Όπως είπα, σέβομαι απόλυτα τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτές που έχει, θα έχει, ακόμα και τις αλλαγές ε, που θέλει στις δικές μας προτάσεις όσον αφορά τον προπολισμό του 2018. Να ξέρετε ότι θα συνεργαστούμε μαζί σας εφόσον ε, καταλήξετε στην τελική σας θέση και την εγκρίνετε επίσημα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εσά ε, προσωπικά κύριε Έτιγκερ προκειμένου να μας βοηθήσετε οι θέσεις μας τελικά να συγκλίνουν και να καταλήξουμε σε ικανοποιητικές συμβιβαστικές λύσεις. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Αρτουή, παρόλο που απουσιάζει, και τον κύριο Μουρεσάν και τον κύριο Άσουερθ που είναι οι για τις ε, επαφές που είχαμε μεταξύ μας και προσβλέπω στη συνέχεια της συνεργασίας μας. Η Ευρώπη στο σύνολό της χρειάζεται ένα προπολογισμό υπεύθυνο που να ταποκρίνεται στις επιθυμίες των ε, πολιτών, ακόμα και αν πρόκειται για κινούμενο στόχο. Και Είμαι βέβαιος ότι με την αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τη δική μας θα μπορέσουμε